Bună Καλώς ήρθατε! Αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια σε όλους τους ευρωβουλευτές που εξελέγησαν ή επανεξελέγησαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα έχουμε την ευκαιρία λοιπόν να συνεργαστούμε στην Επιτροπή Μεταφορών που είναι μια πολύ σημαντική επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και αυτό γιατί μπορούμε να επηρεάσουμε θετικά την ποιότητα ζωής όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας πω ότι σήμερα στην ημερήσια διάταξη έχουμε την εκλογή του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της Επιτροπής μας. Επίσης θέλω να σας ενημερώσω για το ότι η Επιτροπή αυτή θα έχει τέσσερις αντιπροέδρους, όπως είχε και στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν τώρα να ξεκινήσουμε και να περάσουμε στην εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής Μεταφορών ποιο θα είναι ο επόμενο πρόεδρο. Και μετά θα περάσουμε στην εκλογή των αντιπρόεδρων. Είναι σημαντικό να έχουμε το 1 τέταρτο μελών τουλάχιστον παρόντες εδώ για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και στην εκλογή. Είναι εδώ παρόντες, οπότε εντάξει. Θέλω να ρωτήσω τώρα τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων να μου πούνε τι πρόταση έχουν να μας κάνουν για την Προεδρία. Παρακαλώ κύριε Λίκτρετ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για πρώτη φορά έχω συγκινηθεί λίγο που λαμβάνω το λόγο σε αυτή την επιτροπή. Καμιά φορά συμβαίνει και αυτό. Έχω τη μεγάλη χαρά να προτείνω κάποιον για την κοινοβουλευτική μας ομάδα. Υπάρχει εδώ ανάμεσά μας κάποιος ε, ο οποίος ε, ανοίξει αυτούς που έχουν υπηρετήσει μακρόν σε αυτή την, την επιτροπή. Αποτελεί από τους, θεμέλη, τους θεμέλιους λήθους της επιτροπής μας. Είναι ικανότατος, ε, έχει λέγει και είναι ο τέλειος άνθρωπος για την περίπτωση και καθώς από ό,τι φαίνεται μιλά αγγλικά θα μιλήσω κι εγώ τώρα αγγλικά. Θα ήθελα λοιπόν να προτείνω τον κύριο Μπράιαν Σίμψον για την Προεδρία. Domnule Simpson, acceptați candidatura. Κύριε Σίμψον, δέχεστε την υποψηφιότητα αυτή. Ωραία, σημειώνω λοιπόν ότι έχετε κάνει και την δήλωση οικονομικών συμφερόντων. Είσαστε ο μόνος υποψήφιος από ό,τι φαίνεται, οπότε προτείνω να εκλέξουμε τον κύριο Μπράιαν Σίμψον ως πρόεδρο της Επιτροπής μας διαβοής. Συγχαρητήρια. Τώρα, καλό τον πρόεδρο της Επιτροπής Μεταφορών να έρθει παρακαλώ και να αναλάβει την προεδρία της συνεδριάσεως αυτής. Παρακαλώ. an adventure. So the next item is the election of the vice chairs, yeah? Do we do them one at a time, yeah? Yeah. Okay. The Next item on the agenda... Επόμενος είμαι στην ημερήσια διάταξη. Η εκλογή των αντιπροέδρων. Έχουμε τέσσερις αντιπρόεδρους που πρέπει να εκλέξουμε. Πρώτος αντιπρόεδρος, λοιπόν. Υπάρχει υποψήφιος όσον αφορά τη θέση του πρώτου αντιπρόεδρου. Äh, Ο, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σε ευχαριστήσω, να σε συγχαρώ για την εκλογή σου. Δεν ξέρω την ηλικία που απαιτείται για να είναι κανείς ε, πρόεδρος, αλλά το καλό είναι βεβαίως ότι είσαι εδώ πέρα στην αρχή της ε, περίοδου και έχεις αποδείξει επίσης και στο παρελθόν ότι είσαι άνθρωπος του διαλόγου και αυτό είναι θετικό και αυτό ελπίζουμε και για τα επόμενα χρόνια. Σε συγχαίρουμε και εξ ονόματος της ε, ομάδας του ΕΛΚ και επί την ευκαιρία θα ήθελα να προτείνω τον κύριο Ρίκε ως πρώτο αντιπρόεδρο αυτή τη στιγμή, ο οποίος ε, είναι, αν θέλετε, υποψήφιος. Σας ευχαριστώ. Νομίζω πως δεν υπάρχει κάποια υποψηφιότητα για την πρώτη αντιπροεδρία. Οπότε... Ναι, ναι, θα ήθελα μία διευκρίνηση. Εάν ε, μπορούν ε, και τα αναπληρωματικά μέλη να γίνουν αντιπρόεδροι. Νόμιζα ότι δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Ο κανονισμός ε, μήπως άλλαξε μόλις τώρα. The advice I'm getting uh, in is Κοιτάξτε, μου λένε ότι μπορεί να υπάρχει θεσμός, αλλά το ΕΛΚ θα πρέπει να αρνηθεί να έχει ε, τακτικό μέλος στο εγγύς μέλλον. Δεν ξέρω τι σημαίνει το εγγύς μέλλον. Δεν ξέρω, είναι η ειλικρινής απάντηση. Μου λένε ότι είναι δυνατόν όμως. Μάτσες, μπορείς να επιβεβαιώσεις ότι είσαι υποψήφιος. Ναι. Ναι, σύντομα, κύριε Πρόεδρε. Θα πρότεινα να αποδεκτούμε σήμερα την ε, υποψηφιότητα και να το ξεκαθαρίσουμε εσωτερικά μέχρι την επόμενη συνεδρίαση το Σεπτέμβρη, δηλαδή εμείς στο ΕΛΚ. Okay. Καλώς. Ο Μάτιος επιβεβαίωσε την υποψηφιότητα. Το όνομα? Ως πρώτος αντιπρόεδρος ο κύριος Ρίκε. Ο κύριος Ρίκε λοιπόν προτείνεται. Δεν υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες. Δεν υπάρχουν άλλες. Ο κύριος Ρίκε είναι εκεί. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ο κύριος Ρίκε εκλέγεται πρώτος αντιπρόεδρος διαβοής.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 μετά έχουμε εκλογή του δεύτερου αντιπρόεδρου. Ο κ. Μπράντμπορν. Πού είστε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να συγχαρώ, τον, όπως και ο Μάτι Γκρός, σας συγχαίρω για την εκλογή σας. Μπορούμε να βασιστούμε πάνω σας για να ξεκινάμε γέρος τις συνεδριάσεις σε αυτή τη θητεία. Όσον αφορά το κόμμα των Ευρωπαίων Συντηρητικών Μεταρρυθμιστών, Υποψήφιο έχουμε τον κύριο Πίτερ Βαντάλεν, σαν δεύτερο αντιπρόεδρο αυτής της Επιτροπής. Έχουμε υποψηφιότητα λοιπόν του κυρίου Βαντάλεν. Δεν υπάρχει άλλη υποψηφιότητα. Ας εκλέξουμε τον κύριο Βαντάλεν διαβοής λοιπόν. Έχουμε εκλογή τώρα τρίτου αντιπρόεδρο. Κύριε Λάιτουιτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εντάξει, είμαι και λίγο συνηθισμένο στο ρόλο ήδη. Θα... Ως ε, τρίτος... Ε, ως τρίτη ε, αντιπρόεδρο θα, ήθελα θέλαμε να προτείνουμε την κυρία Σιλβία Αντριάννα Τικάου η οποία ήταν και στην ε, προηγούμενη περίοδο. Έχουμε λοιπόν την υποψηφιότητα της κυρίας Τικάου. Δεν υπάρχει άλλη υποψηφιότητα. Εκλέγεται άρα και η κυρία Τικάου διαβοής. Εκλογή τέταρτου αντιπρόεδρου. Κύριε Γκρός. Ναι κύριε Πρόεδρε, εδώ πέρα θα ήθελα να προτείνουμε τον συνάδελφό μου τον κύριο Ντίτερ Κοχ. Έχουμε λοιπόν υποψηφιότητα του κύριου Κοχ. Δεν υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες. Εκλέγεται διαβοής ο κύριος Κοχ. Πριν δώσουμε το λόγο στον κύριο Στέρεξ, να σας υπενθυμίσω ότι η συνεδρίαση μεταδίδεται μέσω του διαδικτύου, μέσω web streaming. Είχε ξεκινήσει το 2008 αυτό. Θα επεκταθεί μετάδοση και θα καλύπτω τη συνεδρίαση όλων των επιτροπών τελικά. Το ανακοινώνω αυτό για τα νέα μέλη κινηματογράφηση γίνεται των ομιλητών όταν πατάτε το μικρόφωνο στρέφεται η κάμερα προς τα εσάς και σας κινηματογραφεί. Αυτές οι συνεδριάσεις συγκροτήσεως σε σώμα κάθε επιτροπής ε, μεταδίδονται μέσω του διαδικτύου. Ήθελα να το ξέρετε. Και υπάρχει ζωντανή κάλυψη συνεπώς της συνεδριάσεως. Συνδέεται αυτόματα λοιπόν η εικόνα με το κουμπί του μικροφώνου. Θέλαμε να το ξέρετε αυτό οτι ώστε να έχετε επίγνωση όταν πατάτε το μικρόφωνο στρέφεται η κάμερα πάνω σας. Αυτά για το web streaming. Ο κ. Στέρξ. Ευχαριστώ. κύριε Πρόεδρε. Με την ε, ομάδα μας των Φιλελευθέρων Δημοκρατών δεν έχουμε υποψήφιο, αλλά θα ήθελα να σας ε, συγχαρώ για την ε, Προεδρία σας και να συγχαρώ και τους άλλους συναδέλφους για την Αντιπροεδρία. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε προβλήματα στην ε, συνεργασία, αν και διαφέρουν οι απόψεις μας. Έχουμε έναν πρόεδρο έμπειρο, ο οποίος τα προηγούμενα χρόνια απέδειξε ότι μπορεί να κάνει και συμβιβασμούς. Αυτά και σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Κράμερ. Ναι. Εδώ. Και εγώ εξ ονόματος των Πρασίνων θα ήθελα να συγχαρώ εσάς κύριε Σίμψον και τους αντιπροέδρους και τις αντιπροέδρους. Έμαθα στην, στον προεκλογικό αγώνα πως ε, η Επιτροπή μας μετά την Επιτροπή Περιβάλλοντος είναι αυτή που νομοθετεί περισσότερο σε ευρωπαϊκό επίπεδο οπότε έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους μας τα επόμενα πέντε χρόνια καθώς χωρίς αλλαγή της ε, πολιτικής μεταφορών δεν θα μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας δεν θα έχουν καμία ελπίδα σε αυτό το πλανήτη. Οπότε πρέπει να μας απασχολήσει αυτό ιδιαίτερα σε αυτή την Επιτροπή και εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους. Ευχαριστώ, Μάικλ. Να σας πω κάτι. Ευχαριστώ όλους όσους πήραν το λόγο για τα καλά σας λόγια. Σας ευχαριστώ για τα συγχαρητήρια που μου δώσατε. Όπως είπα και στην ομάδα μου, είναι πολύ δύσκολο να συνειδητοποιήσω ότι το 1989 θα δώσα το πιο νέο μέλος και το να μπορώ να είμαι πρόεδρος αυτής της Επιτροπής σαν ο μακροβιότερος ε, ευρωβουλευτής, δύσκολο να το συνειδητοποιήσω. Μεγάλο προνόμιο για μένα να είμαι πρόεδρος Επιτροπής Μεταφορών. Όσοι με ξέρετε θα γνωρίζετε ότι όλη την κοινοβουλευτική μου ζωή την πέρασα αυτή την Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι αυτό ήθελα να κάνω. Διότι θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό τον τομέα των μεταφορών και του τουρισμού. Σας παρέχω κάθε διαβεβαίωση και εγγύηση ότι ως πρόεδρος θα είμαι όσο πιο ανοιχτό γίνεται, όσο πιο δίκαιο μπορώ. Θα προσπαθήσω να μιλώ αγγλικά με τα αγγλικά του BBC και όχι με τη συνηθισμένη μου προφορά. Αλλά θα πρέπει να με συγχωρέσετε αν κάποιες στιγμές ξεφεύγω και πάω στην περιοχή του Λάνκασερ και στις ρίζες του Λάνκασερ. Και είμαι περήφανος για τις ρίζες μου. Προσβλέπω σε συνεργασία μαζί σας και είμαι σίγουρος ότι αυτή η Επιτροπή θα συνεχίσει την παράδοση. Δηλαδή συνεργασία, συμφιλίωση, συμβιβασμούς, ούτω ώστε να πετύχουμε τον ευρύτερο, τον γενικότερο στόχο. Διότι όπως ανέφερε και ο Μάικλ, χρειαζόμαστε καλύτερες, αποτελεσματικότερες, ασφαλέστερες μεταφορές τρόπους μεταφορών φιλικότερες προς το περιβάλλον σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσβλέπω στη συνεργασία μαζί σας από τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής και τη συνεργασία η συνεργασία με το προσωπικό ξέρω ότι είναι επιτυχή, διότι ξέρω ότι οι άνθρωποι των μεταφορών, όπω είστε εσεί, θα συμβάλλετε στην επιτυχία μα. Σα ευχαριστώ για τα καλά σα λόγια. Ευχαριστώ για την τιμή και το προνόμιο που μου δώσατε σήμερα προσβλέπω στη συνεργασία μας στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχετε τίποτα για τα διάφορα? Ενέφ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα εννοείται. Μπράιαν, συγχαρητήρια. Σε συγχαίρω από βάθος καρδίας για τη θέση που αναλαμβάνεις. Το μόνο που θα ήθελα στα διάφορα είναι να προτείνω να ασχοληθούμε και πάλι με κάτι για το οποίο είχε δεσμευτεί η Επιτροπή μας πριν από τις εκλογές. Και αυτό ήταν να ζητήσουμε από τον κύριο Πέτερ Χάτσον που ασχολείται με την καταπολέμηση της πειρατείας πλοίων στη Σομαλία να έρθει το φθινόπωρο φαντάζομαι ότι πάλι θα ανέβει η θερμοκρασία στην περιοχή. Καλό θα ήταν να συναντηθούμε μαζί του. Να έρθει και να μας πει και να ακούσουμε και από την Επιτροπή πώς έχουν τα πράγματα περί προϋπολογισμού. Ο αντιπλήρχος λοιπόν αυτός να έρθει να τον ακούσουμε και να δούμε τι μπορεί να κάνει και το Κοινοβούλιο για να βοηθήσει την κατάσταση. Πρόεδρος, ε, να μου επιτρέψεις να πω το εξής. Αυτό που θα κάνω με το έτοιμά σου είναι ότι στη συνάντηση των συντονιστών που θα γίνει, θα το βάλω στην ημερήσια διάταξη, θα το συζητήσουμε και θα δούμε αν η επιθυμία ανανεώνεται και στο καινούριο κοινοβούλιο, ώστε να δούμε και εμείς τι μπορούμε να κάνουμε για την καταπολέμηση της πειρατείας εκεί. Εντάξει, σε ικανοποιεί η αντιμετώπιση αυτή. Καλώ ναι. Καλώς τότε. Άλλο τίποτα? Έχετε τίποτα άλλο? Όχι. Ωραία. Σας υπενθυμίζω μόνο ότι θα συνεδριάσουμε αύριο στις 9 στο κτίριο Γιάν, αίθουσα 4Q1 στις 9, κτίριο Γιάν, αίθουσα 4Q1. Και μετά θα συνεδριάσουν οι συντονιστές. Όσοι είστε συντονιστές θα πρέπει να μείνετε μετά στις 11 για να συνεδριάσουμε παρετέρω. Συμφωνεί. Ωραία, τότε. Είναι Κλείνει η συνεδρία εδώ. Σας ευχαριστώ που ήρθατε και συγχαρητήρια στού στους αντιπρόεδρους για την δικιά τους εκλογή.